Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ευρωβουλευτές, κυρίες και κυρίους. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για τις ερωτήσεις σας, χωρίς καμία εξαίρεση. Προσπάθησα να απαντήσω όσο μπορούσα καλύτερα. Αυτό που μπορώ να σας εγγυθώ είναι ότι έχω τον ενθουσιασμό και έχω και τη θέληση να αναπτύξω περισσότερο τις αρμοδιότητες που μου ανέθεσε ο κύριος Γιούνκερ εφόσον επιβεβαιωθώ στο χαρτοφυλακιό μου. Ειλικρινά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο στην πράσινη ανάπτυξη. Πιστεύω ότι θα είμαστε στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και θα πετύχουμε εμπορικές συμφωνίες οι οποίες δεν θα μας οδηγήσουν σε μετεκατάσταση των βιομηχανιών μας εκτός Ευρώπης και πιστεύω πραγματικά ότι εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε ικανοί να έχουμε ενεργειακά δίκτυα απόλυτα διασυνδεδεμένα και μία εσωτερική αγορά που να λειτουργεί καλά. Γι' αυτό βασίζομαι στο συντονισμό με την Αντιπρόεδρο αλλά και με τους Αντιπροέδρους για την απασχόληση και στη συνεργασία με τους υπόλοιπους επιτρόπους. Πάνω απ' όλα όμως, κυρίες και κύριοι, θέλω να μπορώ να βασιστώ στην συνεργασία μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι απαραίτητο και το ξέρω αυτό από την εμπειρία μου ως Ευρωβουλευτής. 13 χρόνια ήμουνα στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρω ποιες είναι οι επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν λοιπόν έχω την εμπιστοσύνη σας, να ξέρετε ότι θα είμαι επιμονή μου βάσεως στη διάθεσή σας. Θέλω να υπάρχει διαφάνεια απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω και δεσμεύομαι να προχωρήσω σε μελέτες αντικτύπου για κάθε πρότασή μου. Πολύ σοβαρές μελέτες και πολύ αυστηρές και για τις οικονομικές επιπτώσεις και για τις κοινωνικές επιπτώσεις και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θέλω επίσης η διαβούλευση με τους πολίτες να είναι σε μόνιμη βάση και να είναι σοβαρή η διαβούλευση αυτή. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργάζεται μαζί μου από την αρχή της κάθε πρωτοβουλίας. Έτσι, χέρι-χέρι θα προχωρήσουμε στις σημαντικές δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβουμε, διότι οι στόχοι μας είναι περίπλοκοι. Πρέπει να έχουμε ηγετική θέση στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να μιλάμε με μία μόνο φωνή. Πρέπει να διαπραγματευόμαστε με μία φωνή όταν μιλάμε για την αγορά εκπομπών. Πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι παραπάνω από 28 χώρες μαζί. Και έχω τη στήριξη δύο ε, γενικών διευθύνσεων που τις γνωρίζετε πολύ καλά. Η Επιτροπή Ήτρε συνεργάζεται με τη μία και η Επιτροπή Ένβη με την άλλη. Υπάρχουν εξαίρετοι αξιωματούχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν τις καλύτερες δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα καλύτερα προσόντα. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε συντονισμένα. Ξέρω ότι ορισμένοι από εσά έχουν ε, επιφυλάξεις όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο αυτό. Αλλά πιστεύω ότι αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για όλους, με επιλογές καλά ισορροπημένες, φιλόδοξες πάντα. Και εννοείται, είμαι σίγουρος ότι αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά, θα δώσουμε και απάντηση στα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επόμενες γενιές το αξίζουν. Αξίζουν ένα περιβάλλον καλό, βιοπικιλότητα, δεν πρέπει να θέσουμε τις επόμενες γενιές σε κίνδυνο όσον αφορά τα θέματα αυτά. Τα 5 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη επίσης απαιτούν μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θέλουν οικονομική ανάπτυξη. Θέλουν οι περιβαλλοντικές μας προδιαγραφές να συνοδεύονται από την ανάπτυξη αυτή. Είναι μια ισορροπία δύσκολο να επιτευχθεί. Δεν είναι εύκολη. Και το ξέρω. Γι' αυτό και δεσμεύομαι απέναντί σας να προχωρήσω προς τους στόχους αυτούς με τη δικιά σας συνεργασία, με τη συνεργασία όλων. Είμαι συνεπώς στη διάθεσή σας εφόσον ε, έχω την εμπιστοσύνη σας και συγχρόνως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας και τις ερωτήσεις σας σε αυτή την ακρόαση. Uh, Σας ευχαριστούμε κύριε υποψήφια επίτροπε. Έχουμε τηρήσει πιστά το χρόνο μας και κάποιες πληροφορίες. Θα δώσω το λόγο στον Συμπρόεδρο Λαβία για να μας ενημερώσει για τα διαδικαστικά, ιδιαίτερα για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ Γέζη. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές, τον προτινόμενο επίτροπο, για τις ερωτήσεις και απαντήσεις και να ενημερώσω τους συντονιστές της Επιτροπής Περιβάλλοντος ότι η συνεδρίασή μας για την αξιολόγηση, την κοινή αξιολόγηση θα γίνει 10 με 11.30 αύριο το πρωί. Ενώ στις 11.30 με 12.30 θα έχουμε την κοινή συνεδρίαση των συντονιστών των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας, MVK για να αποφασίσουμε. Ευχαριστώ και ξαναδίνω το λόγο στον πρόεδρο Μπούζεκ. Τώρα, για τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Ξέρετε οι συντονιστές πότε θα συνεδριάσουμε για την αξιολόγηση. Το πιο σημαντικό όμως είναι η επόμενή μας ακρόαση. Στη μιάμιση, αύριο, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ε, Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη, τους συμπολίτες μας που μας παρακολουθούν απευθείας ε, μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους έλαβα μέρος στην ακρόαση και ιδιαίτερα τον υποψήφιο επίτροπο. Καληνύχτα σας.